Θα ήθελα λοιπόν να σας επισημάνω ότι στον τρίτο γύρο ισχύει πλέον η απλή πλειοψηφία. Ο κύριος Λούκα. Λούκε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μας εξηγήσετε πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν άκυρα ψηφοδέλτια. Πρόεδρο, μπορείτε να ψηφίσετε και το μηχάνημα καταγράφει την ψηφοφορία σας και μετά μπορείτε όμως να τα σβήσετε ε, και αυτό θεωρείται άκυρο. Δηλαδή έχετε τη δυνατότητα να αρνηθείτε να ψηφίσετε. Πατάτε μία φορά και μετά σβήνετε όλα τα ονόματα. Στην περίπτωση αυτή είναι άκυρη η ψήφο σας. Αν θέλετε αυτό είναι το λευκό ε, ψηφοδέλτιο ε, κάτι το οποίο και στην ψηφοφορία διαλληλογραφίας θεωρείται άκυρο. Πάμε τώρα στον επόμενο γύρο και σας παρακαλώ πολύ να περάσετε τα ονόματα και όταν θα είναι ε, δυνατόν να ανοίξει η ψηφοφορία παρακαλώ πολύ να με ειδοποιήσετε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Έκανα ένα λάθος ε, που αφορά στον κύριο Ρέιντεν. Ρέν. Ε, τον κύριο Ρέν, με συγχωρείτε. Είχε 304 ψήφους και όχι 384. Κατόπιν ζούτο ο κύριος Ρέν δεν εξελέγει, άρα δηλαδή αναφέρεται τώρα σε αυτό το γύρο ως υποψήφιος. Δεν ξέρω γιατί έκανα λάθος, ε, μάλλον διάβασα λάθος αριθμό, αλλά κύριε ε, Ρεν, σας ζητώ συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ, θα πρέπει να υποβάλλετε την υποψηφιότητα για άλλη μια φορά στον τρίτο γύρο. Λοιπόν, τώρα όμως μπορούμε να ψηφίσουμε. Κύριε Γκασπάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Πάμε τώρα στον τρίτο γύρο. Βλέπετε τα ονόματα και τώρα ψηφίζουμε για τρίτη φορά, στον τρίτο γύρο. Haben Ψηφίσατε όλοι παρακαλώ. Μήπως υπάρχει κάποιος που ψηφίζει ακόμα. Από ό,τι βλέπω όχι. Κατόπιν τούτου κλείνει η ψηφοφορία. abgegebene Stimmen. Λοιπόν, ψήφισαν. 306. 690 έγκυρα, άκυρα 16. 346 είναι απαιτούμενη πλειοψηφία, 346 ψήφοι. Η απόλυτη πλειοψηφία, αλλά τώρα αρκεί η απλή πλειοψηφία. 377 Ρέιν, Λάμπστορφ, 365 Λούνατσεκ, 319, Παπαδημούλης 302, Τσανέτσκι 284, Καστάλντο 110. Λοιπόν, ως εκ τούτου εξελέγησαν Ρέν, Λαμπστόφ, Λούνατσεκ, Παπαδημούλης και Τσανέτσκι. Υπάρχει κάποιος που δεν αποδέχεται την εκλογή του. Από ό,τι βλέπω όχι, την αποδέχονται όλοι, Συγχαρώ, συγχαίρω λοιπόν όλους και ως εκ τούτου εξελέγει και το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τώρα την ε, εκλογή των κοσμητόρων. Προτείνω μέχρι αύριο το πρωί στις 10 να ισχύει προθεσμία για την υποβολή υποψηφιωτήτων. Τετάρτη, 10 η ώρα το πρωί, καταληκτική ημερομηνία και παρακαλώ να κατατεθούν υποψηφιότητες στην αίθουσα R00101 και να παραδώσουν την υποψηφιότητα στα χέρια του Γενικού Γραμματέα. Η συνεδρίαση διακόπτεται και συνεχίζουμε αύριο το πρωί στις 9.